Ε, ένα αίτημα για διορισμό σε επιτροπή του Μάρκου Πρέτσερ στην ε, Επιτροπή Μέτρησης Εκπομπών Ρήπων Αυτοκινήτων. Αυτό θα καταχωρηθεί στα πρακτικά και με την έγκριση, αν δεν υπάρξει ένσταση γι' αυτό θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται αυτός ο διορισμός.